τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε μια τόσο δύσκολη περίοδο οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαβία. Και τώρα ολοκληρώνεται το σημείο αυτό, το οποίο θα ψηφιστεί αύριο στις 12. Και παίρνουμε στην κοινή συζήτηση τώρα για τον τομέα του κακάο, στη σύσταση του κυρίου Μορέιρα, για τη Διεθνή Σύμβαση για το Κακάο το 2010 και την δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο. Το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά ο κύριος Μορέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ Θέλω να θέσω ευθύ εξ αρχή τη συζήτηση δύο θέματα τα οποία είναι αλληλένδετα αν και διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα η Διεθνή Σύμβαση για το Κακάο για το 2010, συμφωνία για την οποία ζήτησα την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεύτερον ένα ψήφισμα, σχέδιο ψηφίσματος για την παιδική εργασία στον τομέα του κακάο. Είμαι ο αρμόδιος εισηγητής της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και για τη συμφωνία και ένας από τους συντάκτες του σχεδίου ψηφίσματος που η ίδια αυτή επιτροπή θα υποβάλει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Ως προς το πρώτο θέμα, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε ομόφωνα το να δώσει το Ευρωκοινοβούλιο πράσινο φως ώστε να συνευθεί η Διεθνή Σύμβαση για το Κακάο για το 2010. Για τρει θεμελιώδει λόγου. Πρώτον, η συμφωνία αυτή ενισχύει την δυνατότητα διακρατική συνεργασία στον τομέα του Κακάο ώστε να υλοποιηθούν στον ίδιο αυτό τομέα οι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί. Επίση, η συμφωνία επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια στην μορφή που λειτουργεί ο οργανισμός για το ΑΚΑΟ, καθώς και το πώς συμμετέχουν οι οργανισμοί του κοινωνίας των πολιτών στην όλο αυτό το τομέα. Και επίσης, κατά τρίτον, γιατί υπάρχουν νέα διατάξεις που μπορούν να προωθήσουν τις καλύτερες εργατικές σχέσεις και την βιώσιμη οικονομία στον τομέα του ΚΑΚΑΟ. Η συμφωνία απαιτεί από τα συμβαλόμενα μέρη να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας με ε, κανόνες, τρόπους που διεθνώς να αναργωνίζονται από τη Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Επίσης, ε, παροτρύνει τις συμβαλόμενα μέρη να προωθήσουν την βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας του κακάου και να εφαρμόσουν προγράμματα τα οποία επιδιώκουν ακριβώς τους στόχους αυτούς. Ως προς τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κακάου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχει αυξημένη ευθύνη ώστε να βεβαιωθεί ότι η παραγωγή και η εκμετάλλευση των φυτών κακάο γίνονται κατά τον τρόπο τον, πιο, πλέον διαφανή και βιώσιμο. Ο τομέας του κακάο είναι ο διεθνή μάλλον οργανισμό του κακάο είναι μάλλον ο μεγαλύτερο σύμμαχό μα για να μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου αυτού. Τώρα, ω προ το δεύτερο ψήφισμα που ανέφερα. Η παιδική εργασία στον τομέα του κακάο με τι ε, ε, εξαγωγέ είναι πολύ σημαντική διάσταση όταν θέλουμε να δώσουμε την έγκρισή μας, μάλιστα στη Διεθνή Συμφωνία για το Κακάο. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο προτείναμε και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου το δέχτηκε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, όπου εκφράζονται κάποιες από τις μέρημνές μας σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται η παιδική εργασία στις φοιτίες κακάο, ιδίω στη Δυτική Αφρική. Αυτό ε, αφορά και τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Όλοι ευαισθητοποιούνται για το θέμα αυτό, όπως και οι πολιτικοί ευθύνοντες. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία υπήρξε έντονη κινητοποίηση της διεθνούς βιομηχανίας του κακάο, ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των συμβαλωμένων και των ενδιαφερομένων μερών, όπως οι διεθνείς ε, θεσμοί, ε, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να περιοριστεί η παιδική εργασία στον τομέα του κακάο. Βεβαίω, πολλά απομένουν να γίνουν. Διότι τα παιδιά που εργάζονται στον τομέα του κακάο είναι εκτεθειμένα σε κινδύνου, ιδίω στον τομέα τη υγεία. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, βεβαίω, για το τι διαστάσει έχει ακριβώ το φαινόμενο. Μιλάμε όμω για δεκάδε ή εκατοντάδε ενδεχομένω εκατομμύρια παιδιών. Ε, και βεβαίω αυτό αρκεί για να μα ε, ανησυχεί και για να μην αφιστούμε προσπαθειών ώστε να περιορίσουμε ε, την εργασία των παιδιών που είναι ένα από τα πλέον επιβαρυντικά στοιχεία για τον τομέα του κακάου. Η παιδική εργασία είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιγόντω ε, μεταξύ των ε, ηθινών των, ε, πολιτικών αποφάσεων, αυτών που λαμβάνουν πολιτικέ αποφάσει, των υπευθύνων τη κοινωνία πολιτών και των κυβερνητικών οργανώσεων και των θεσμικών οργανών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, να έχουμε συγκεκριμένε προτάσει στα χέρια μα ικανοποιητικέ για το πώ προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναχαιτήσει, να ανταποκριθεί μάλλον στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μορέιρα. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Πίπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα ξεκινώντα να ευχαριστώ τον κύριο Μορέιρα και την Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου για τις προτάσεις προς το Κοινοβούλιο, ώστε να ε, εγκρίνει την, να δώσει συμφωνή γνώμη για την συμφωνία αυτή, τη Διεθνή Συμφωνία. Είναι μια νέα συμφωνία και συμφωνεί το Κοινοβούλιο ότι αποτελεί μια καλή βάση για την προαγωγή της διεθνούς συνεργασία στον χώρο του κακάου και θα συμβάλλει στην ενίσχυση των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών παράγων κακάου. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία τίνει προς την εξασφάλιση δίκαιων τιμών, προς όφελο τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή, προάγει όμως ταυτόχρονα και της, ε, την ισότιμη ανταπόδοση της παραγωγής και την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα του κακάου. Μην ξεχνάμε ότι οι χώρες που παράγουν κακάο σε μεγάλο βαθμό είναι και αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές του κόσμου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, έχει σαφώς ε, ευθύνη για να προαγάγει ένα δίκαιο εμπόριο κακάο στις χώρες αυτές. Με αυτή την ευθύνη λοιπόν υπόψη αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα του, της παιδικής εργασίας αποτελεί μια από τις κύριες προκλήσεις Διαφιλονικούμενο σημείο είναι ότι κατά την άποψή μας αυτή η ιδέα είναι απαράδεκτη, είναι αποτρόπαια, ενώ σε άλλες ε, κουλτούρες και πολιτισμούς είναι αποδεκτή πρακτική. Έτσι λοιπόν ε, και όπως λένε διάφοροι οργανισμοί μεταξύ των οποίων και ο Παγκόσμιος, ε, το Παγκόσμιο Ίδρυμα για το Κακάο ε, μπορεί να αποτελέσει η λύση αυτή μια καλή βάση για την πρόοδο στο χώρο της, του εμπορίου στο κακάο. Εμείς όμως λέμε ότι η παιδική εργασία δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο του κακάο, αφορά και επηρεάζει σχεδόν όλες τις χώρες εταίρους, αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους τα δικαιώματα των παιδιών. Ξέρετε ότι έχουν ε, παγιωθεί μέσα στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καθήκον μας είναι να προαγάγουμε τα δικαιώματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ρητά στρατευμένη στο στόχο αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη στην ε, απάλληψη κάθε μορφής παιδικής εργασίας ανά τον κόσμο και στην διασφάλιση ότι η εκπαίδευση του παιδιού δεν θα θυσιαστεί στο βωμό της ανάγκης για εργασία. Η φυσική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού δεν θα επηρεαστεί από την παιδική εργασία. Σε διεθνές επίπεδο και υπό το άρθρο 32 της ε, Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται ότι τα, τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασίας από την οικονομική εκμετάλλευση και την παιδική εργασία. Πριν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανελειμμένως εξέφρασε την βαθύτατη λύπη της για το γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας συμπεριλαμβανομένης και της ε, Σύμβασης 182 ε, που κυρώθηκε σχεδόν από όλες τις χώρες και που απαγορεύει την εργασία των παιδιών. Υπάρχουν ακόμη πολλές χώρες οι οποίες ε, αναπτύσσουν δραστηριότητες που εντάσσονται στον χώρο, στον ορισμό μάλλον του Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας για την παιδική εργασία. 120 εκατομμύρια παιδιά είναι στον κόσμο σήμερα αυτά που εργάζονται, 30% των παιδιών στην υποσαχάρια Αφρική συγκεκριμένα. Αυτά όλα πρέπει να μας οδηγήσουν σε σκέψεις και χαίρομαι για τις προτάσεις του κύριου Μορέιρα που υποστηρίζουν πολλοί βουλευτέ του Κοινοβουλίου και, στη σημασία, και τη σημασία που αποδίδουν στο θέμα αυτό. Το θέμα όμω είναι περίπλοκο. Στις αναπτυσσόμενες χώρες και ειδικότερα στον χώρο του κακάο, το πρόβλημα της παιδικής εργασίας δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένο. Μια ολιστική προσέγγιση πρέπει να αντιμετωπίζει και άλλα ζητήματα που απορρέουν από το πρόβλημα της φτώχειας και της ως εκ τούτου ανάγκης να δουλέψουν τα παιδιά, ακόμα και της διακίνησης παιδιών, εμπορίας παιδιών για να εργαστούν στον χώρο αυτό. 9% των ε, φοιτιών ε, κακάο ανήκουν σε μικρές επιχειρήσεις, οικογένειε, που αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις και που μερικές φορές ε, απέχουν 40 χιλιόμετρα από τον εγκύτερο δρόμο και δεν έχουν καμία υποδομή στη θέση τους. Έτσι λοιπόν από αυτές τις συνθήκες βεβαίως και θα δουλέψουν στο Ινφιτία την οικογενειακή τα παιδιά. Για να στηριχθούν λοιπόν οι κοινότητες ώστε να προσφέρουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες δεν θα επιχωρούν πλέον τα παιδιά να εργάζονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας και των πολιτικών που εφαρμόζουν στο μέα αυτών συνεχίζει τις προσπάθειές της. Έχουμε μια στράτευση να λάβει και έχουμε περιγράψει στο πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2010 και, τις, ε, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2010 για, τον περιορισμό της, ε, για την εξάλληψη παιδικής εργασίας και κάνουμε διαρκείς και σταθερές προσπάθειες στο τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε θεσπίσει ε, μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση συνεργαζόμενη με τους αρμόδιους και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και σώματα. Η χώρες της Δυτικής Αφρικής ε, μπορούν να, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό μόνες τους μέσω της συνεργασίας με τη βελτίωση των υποδομών, με τη βελτίωση των γεωργικών μεθόδων, με ε, καλύτερες, ε, καλύτερη επιθεώρηση εργασίας, καλύτερη οργάνωση αγοράς, παραδείγματι. Και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι πιστεύω ακράτα πως η ενός παιδιού είναι στο θρανείο του σχολείου του και όχι στην φοιτεία και τη γεωργική εκμετάλλευση. Η εκρίζωση όμω τη φτώχεια πρέπει να είναι ο πρώτο στόχο τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, για να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τη ρίζα του κακού τη παιδική εργασία στην Δυτική Αφρική αλλά και σε όλε τι αναπτυσσόμενε χώρε. Με ιδιαίτερη λοιπόν ευγνωμοσύνη σημειώνω προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την διαπίστωση ότι το θέμα αυτό το έχει θέσει υψηλά στο πρόγραμμά του και ως συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει το καθήκον αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Από το ΕΛΚ, η κυρία Γκέστιγκε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απευθυνθώ στον εισηγητή και τους συναδέλφου των άλλων ομάδων και να τους ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Νομίζω με την έκθεση αυτή και κυρίως με το ψήφισμα καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό. Η νέα συμφωνία βεβαίως είναι σημαντικό βήμα ε, ανάμεσα στις χώρες συνεργασίας για τις χώρες που παράγουν και τις χώρες που καταναλώνουν κακάο. Θα πρέπει να έχουν μια δυνατότητα προγραμματισμού οι οικογένειες των καλλιεργητών κακάο και να υπάρχει και μια ασφάλεια ε, καταπολέμηση ταυτόχρονα της εργασίας που εκμεταλλεύεται τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς έχουμε ευθύνη στο μέλλον ε, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύσει αυτές να εξελιχθούν προς ένα δίκαιο ε, τρόπο καλλιέργειας. Ε, ασχολούμαστε με την καταναγκαστική εργασία των παιδιών στο ψήφισμά μας και πέρα από πολιτικές ομάδες καταφέραμε να συμφωνήσουμε. Το θέμα είναι πώς ορίζεται η παιδική εργασία, γιατί δεν είναι κάθε παιδική εργασία ούτε επικίνδυνη ούτε εκμετάλλευση. Αυτό φαίνεται και στις κύριες ε, παραγωγούς κακάο. Τελικά ε, είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και εκεί βοηθούν τα παιδιά τους γονείς τους. Σημαντικό είναι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση τα παιδιά και να αναπτύσσονται γενικά. Αυτό που μας ε, προβληματίζει είναι ε, καταστάσεις καταναγκαστικής εργασίας των παιδιών, εκμετάλλευσης και συνθήκων που απειλούν την υγεία τους γιατί είναι επικίνδυνες. Και γι' αυτό σας λέγω ότι είναι ισόρροπο το ψήφισμα και οποιαδήποτε αλλαγή είναι περίτη. Και θα χαιρόμουν αν ο εισηγητής καταφέρει και μεταφέρει και στην Ολομέλεια την καλή συνεργασία και το πνεύμα που επικράτησε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Για ένα λεπτό η κυρία Παντία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι, καταρχά θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μορέιρα για την καταπληκτική του εργασία και του ψηφίσματο και για τη συμφωνία. Αυτή είναι η Διεθνή Συμφωνία για το Κακάο που θα ψηφίσουμε αύριο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι συμπεριλαμβάνει μέτρα που βελτιώνουν την προηγούμενη συμφωνία. Μέτρα όπω είναι η ανάπτυξη των παραγωγικών οικονομιών, οι σωστέ τιμέ και δίκαιε και για παραγωγού και για καταναλωτέ και ένα αηφόρο πλαίσιο και ω προ το περιβάλλον αλλά και ω την κοινωνική πτυχή. Και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό το πλαίσιο εδώ το κοινωνικό ε, επιμένει το ψήφισμα που συνοδεύει αυτή τη συμφωνία και που επίσης αύριο θα ψηφίσουμε. Και πιστεύω ότι το γεγονός ότι επιμένει κυρίως στην εξάλληψη της παιδικής εργασίας είναι μεγάλο επίτευγμα και κατάκτηση. Είναι από τα προβλήματα που έχουμε, το είπε και ο Επίτροπος, εδώ και χρόνο προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, αλλά το γεγονός είναι ότι ε, οι αριθμοί που μας έδωσε 124 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο εργάζονται. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα χαροποιό. Θα πρέπει να δοθεί αυτή η μάχη παντού, σε πολλά μέτωπα. Είναι ε, ζωτική σημασίας θα πρέπει να κυρωθεί υποχρεωτικά η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού από όλε τι χώρε. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και δεν ε, ακούστηκε εδώ, να γίνει πρόοδο στην έρευνα και την ανάπτυξη για να έχουμε τεχνικέ καλλιέργειας και συγκομιδή του κακάο που να μην ε, υποχρεώνουν τα παιδιά να εργάζονται. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο ευρωπαϊκό κανόνα και προδιαγραφή για την αηφορία και την ε, η χνηλασιμότητα των προϊόντων. Θα ήθελα παρακαλώ τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Αμπαντία, λέει ο Πρόεδρος. Εντάξει, ικανοποιηθήκατε, αλλά ένα λεπτό είχατε. Μην το ξεχαράτε ότι σας έχω κάνει χάρη. Ε, λοιπόν, από τους φιλελευθέρους και δημοκράτες για δύο λεπτά ο κύριο Ρινάλντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η αγορά το κακάο είναι παρά, κάτι το παράδοξο, διότι είναι τόσο γλυκό το τελικό προϊόν, αλλά σχεδόν καταραμένες οι πηγές του προϊόντος αυτού. Η αρχή του εμπορίου του κακάου, γύρω στο 1500, με τη χρήση εμπορικών πλοίων ε, βασιζόταν στην, ε, στα σκλαβοβάζαρα και την δεν μπορεί δούλων για να χρηματοδοτήσει την ε, παραγωγή του προϊόντος αυτού. Στην Γκάνα με 60% της παγκόσμιας παραγωγής είναι τεράστιος ο ρόλος των παιδιών στην ε, στην παραγωγή του προϊόντος αυτού. Ήδη την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην ακτή του Ελεφαντοστού για την ετήσια συνδιάσκεψη των ε, χωρών της Αφρικής που παράγουν κακάο με την παρουσία μη κυβερνητικών οργανώσεων που προσπαθεί να καταπολεμήσει την παιδική εργασία στις περιοχές που παράγουν κακάο. Ο πρόεδρος Κακάο έδωσε αρχή στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας ε, με την ε, σύμβαση ε, που θα υπογραφεί αυτή. Όμως εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, ανάληψη κοινωνικών ευθυνών στον τομέα του Κακάου, διότι για αυτόν τον λόγο ακριβώς χρησιμοποιούνται οι δηλητηριασμένε μέθοδοι για τους εργαζομένους επειδή δεν υπάρχει ανταντικοποίηση, εκβιομηχάνηση της παραγωγής του κακάου. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερο διαφανής ε, ε, παραγωγή σαφέστερη, χωρίς να υπάρχει εκμετάλλευση των εργαζομένων. Για τις ε, εισάγουσες χώρες που ανήκουν και στο Διεθνή Οργανισμό Κακάο υπάρχουν ειδικέ ευθύνε. Τη σωστή εφαρμογή τη συμφωνία και προκειμένου να γίνει αυτός, αυτή η συμφωνία ένα εργαλείο, ώστε να καταπολεμήσουμε τι ε, μεγάλε αδικίες που υπάρχουν στον χώρο τη παραγωγή του κακάο. Αλλά δεν αρκεί μόνο της η σύμβαση. Θα πρέπει και οι καταναλωτές να έχουν καλύτερη επίγνωση ε, του τι συμβαίνει στον τομέα του Κακάου, να έχουν επίγνωση ότι πρέπει να καταφεύγουν στα προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί σε συνθήκες ε, ισότιμου ανταγωνισμού χωρίς παιδική εκμετάλλευση και χωρίς ε, παιδική εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε τόνο στι ε, όθησε τη προσπάθεια αυτέ που μέχρι τώρα έχουν παραμείνει προσπάθειε ιδιωτών. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματο τη ομάδα του, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Στά. Συνάδελφοι, πρόεδρε, επίτροπε. 70% παγκόσμια παραγωγής κακάο είναι από την Κάνα και την ακτή ελεφαντοστού. 80% εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Δυτική Αφρική. Γνωρίζουμε όλοι τις αναρρύθμιτες εκθέσεις για την παιδική εργασία και πραγματικά είναι ανησυχητικό αυτό. Στην Ένωση θα πρέπει ε, να ξέρουμε ότι έχουμε και τη μεγαλύτερη βιομηχανία σοκολάτας ε, είναι κάτι σοβαρό και σημαντικό και θα πρέπει να επικρατούν εκεί καλές συνθήκες και κοινωνικές και οικονομικές. Και είναι καλό που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και συμπεριλαμβάνουμε και την παιδική εργασία. Καλό είναι το ψήφισμα του συναδέλφου Μορέιρα. Και δίνει έναν από τους δύο τρόπους που μπορούμε να αποφύγουμε ε, την παιδική εργασία. Ο ένας τρόπος είναι πραγματικά να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία, ανταλλαγή know-how, τεχνογνωσίας, ο καθένας να συνεργάζεται σωστά και ο τομέας της διανομής να μην βρίσκουν διέξοδο στην αγορά προϊόντα από φοιτίε που απασχολούν παιδιά. Αλλά ο άλλος δρόμος είναι οι καλέ και σωστέ διεθνεί τιμέ. Και η σημερινή συμφωνία θα πρέπει να βοηθήσει προ αυτή την κατεύθυνση ε, πραγματικά με σθένο και ε, όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Γιατί όταν είναι σωστέ οι τιμέ αποφεύγουμε την παιδική εργασία. Όταν είναι χαμηλέ οι τιμέ, επικρατεί η ένδυα που δεν οδηγεί στη σωστή εργασία. Να φροντίσουμε λοιπόν για δίκαιε και σωστέ τιμέ, Αυτό είναι απόλυτο και πάρα πολύ απαραίτητο σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα για ένα λεπτό ο κύριος Σόλτς. Χωρίς μικρόφωνο. Ε, αναφερόμαστε στην παιδική εργασία. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη φορά να το ε, καταδικάζει ε, ως ε, φτηνή πηγή εργασίας. Ε, όμως ε, δεν ήταν ε, αξιοπρεπή η συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επιτροπή. Εάν θα πρέπει να καταδικάσουμε μόνο την καταναγκαστική εργασία των παιδιών ή γενικά την παιδική εργασία σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Προσοχή κύριε Στέρντ, κινδυνεύουμε να οπισθοδρομήσουμε. Ε, η ε, παράγραφος η αιτιολογική σκέψη μάλλον ε ωρεοποιεί την κατάσταση ε, των παιδιών. Δεν έχουν ευκαιρίες στη μόρφωση και στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Και κυρία Κιώστιγκερ και οι συνάδελφοι του ΕΛΚ στην αιτιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑ καταφέρατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κλείσει τα μάτια του μπροστά στο γεγονό ότι γίνεται εμπόριο παιδιών στι φοιτίε, ιδιαίτερα στην Κάνα και στην ακτή ε, Ελεφαντοστού. Είναι ικτρή η πραγματικότητα. Κοιτάξτε το ντοκιμαντέρ ε, «Βρώμικη σοκολάτα». Ένα παιδί κοστίζει 230 ευρώ. Τα φέρνουν από το Μαλί, από όπου τα απαγάγουν. Η διεθνή Οργάνωση Εργασίας ε, έχει μετρήσει πάνω από 12.000 παιδιά στι φοιτίε τη ακτή Ελεφαντοστού που δεν έχουν συγγενεί την άλλη φορά, κύριε Επίτροπε και συνάδελφοι, που θα φάτε σοκολάτα, για σκεφτείτε ποια παιδική μοίρα σας έχει δώσει αυτή την απόλαυση. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό από τους μία εγγεγραμμένους τώρα το λόγιο έχει ο κύριος Μέλτσερ. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι ο τομέα του κακάου βρίσκεται πίεση Είναι αυξημένη η ζήτηση κυρίως από την Ασία για το κακάο και ταυτόχρονα περιορισμένη συγκομιδή τα τελευταία χρόνια. Ένα εκατομμύριο τόνι κακάο λιγότερο από ό,τι χρειάζεται διατίθεται στην αγορά αυτή την εποχή τα τελευταία χρόνια. Και ιδιαίτερα η κυβέρνηση της ακτής του ελεφατοστού θα πρέπει να κοιτάξει τους όρους υπό τους οποίους παράγει το κακάο. Το 2012-2013 η συγκομιδή του κακάο ε, πολίθηκε πρόωρα σε κρυφούς πληστηριασμούς, ε, παράνομα δηλαδή ε, διατέθηκε αυτή η συγκομιδή. Μέσα από συνθήκες παράδεκτης εργασίας παιδιών παράγονται αυτά τα προϊόντα και αν θέλουμε να καταστήλουμε αυτή τη ε, μέθοδο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής σοκολάτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξει στάση. Θα πρέπει να επιδιώξουμε ένα πιστοποιημένο ε, και βιώσιμο σύστημα παραγωγής κακάο. Ευχαριστώ πολύ και τώρα οι επόμενοι ομιλητές για ένα μισό λεπτό ο κύριος Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, στο θέμα αυτό και πολλοί το υπογράμμισαν σήμερα, Βρισκόμαστε ενώπιον ενό διλήμματο ότι δηλαδή απορρίπτουμε όλοι επί τη αρχή την ε, παιδική εργασία και εγώ ω πατέρα τεσσάρων παιδιών αισθάνομαι ε, βαριά στη συνείδησή μου ε, τη γνώση του πόσα παιδιά πρέπει να δουλέψουν για να πιούν τα δικά μου το πρωί, στο πρωινό τους ένα φλιτζάνι κακάο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ελάχιστε προδιαγραφές επιβίωσης για τα κράτη αυτά και τις υποδομές που χρειάζονται όπως σχολεία, όπως υποδομές, όπως κοινωνικά συστήματα. Το δίλημα λοιπόν το οποίο αντιμετωπίζουμε ότι αν δεν αναπτύξουμε τι εμπορικέ συναλλαγές με τα κράτη αυτά, εάν δεν αγοράσουμε τα προϊόντα τους δεν θα μπορούν να αναπτύξουν τις, ε, τις υποδομές αυτές που χρειάζονται. Αλλά από την άλλη αν αναπτύξουμε τις εμπορικές συναλλαγές ίσως να παραγνωρίσουν τις ε, υποχρεώσεις τους για τη ρίση των βασικών αρχών. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστώ τους αδέλφους ε, που συζήτησαν το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η συμφωνία είναι μια καλή λύση, ένας καλός δρόμος. Κοιτάμε δηλαδή ανοιχτά το θέμα των εμπορικών συναλλαγών με τα κράτη αυτά, των εμπορικών συμβάζων και σχέσεων. Λέμε όμως ταυτόχρονα στα κράτη αυτά ότι θέλουμε να τα βοηθήσουμε να ξεφύγουν από, την, από το δίλημα αυτό. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να έχουμε ένα καλό, μια καλή ε, σοκολάτα ή ένα καλό κακάο, αλλά και καλό μέλλον για τα παιδιά αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούστα. Κύριε Πίτροπε, συνάδελφοι, εδώ η στόχοι τη συμφωνία ε, είναι στόχοι που μπορούμε να συμμεριστούμε και πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία αυτή. Όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που διατρέχει όλο αυτό το τομέα. Εμπόριο που θα βελτιώσει τι συνθήκε τη παραγωγή, ναι, με, με σωστέ τιμέ ε, βεβαίω, αλλά θα πρέπει να μην επιδίων να επιδιώξουμε και βελτίωση των συνθήκων ε, των 5,5 εκατομμυρίων καλλιεργητών και 14 εκατομμυρίων εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα του κακάου. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να πιέσουμε τους, ε, επεξεργαστέ και παρασκευαστές να καταπολεμήσουν, να αναχαιτήσουν την εκμετάλλευση των... της των παιδιών ε, και να υπάρξει ισότιμο, ισό... αγορά με ισότιμους όρους στον τομέα του κακάο. Βιώσιμη αγορά. Ευχαριστούμε. Κύριε Σούστα. Για ένα λεπτό, κύριος Κούτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μην ξεχνάμε ότι 158 εκατομμύρια παιδιών ε, κάτω των 15 απασχολούνται στο τομέα του κακάο. Ένα στα έξι παιδιά ε, που θα έπρεπε να πηγαίνουν στο σχολείο. Εκατομμύρια είναι τα παιδιά που εργάζονται στον τομέα αυτό και των οποίων πλήττεται η υγεία λόγω των χημικών ουσιών ε, ε, χιλιάδε παιδιά εργάζονται σε δυσχερεί ε, συνθήκε στι φυτίε του κακάου και πολλά από αυτά είναι θύματα εμπορία. Οι εμπορικέ τιμέ ε, του κακάου, οι τιμέ τη αγορά, πιέζουν του καλλιεργητέ να καταφύγουν στην παιδική εργασία. Αυτό έχει προφανώ σοβαρότατε συνέπειε για την υγεία των παιδιών και για τη σχολική τους εκπαίδευση. Νομίζω ότι η πρόσβαση στην παιδεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και να δοθεί τέρμα στην εκμετάλλευση των παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να πιέσει τα κράτη που καταφεύγουν στην παιδική εργασία. Να σας θυμίσω ότι μπορούμε να αναστείλουμε τις εμπορικές μας συμφωνίες στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, εάν το θέλουμε. Επίσης, όλες οι συμφωνίες μας με τις θα πρέπει να έχουν διατάξεις ό,τι αφορά την βελτίωση σε των συνθηκών εργασία των παιδιών. Ευχαριστώ κύριε Κούτα. Για ένα λεπτό κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υποστηρίζω βεβαίω ε, τη Διεθνή Συμφωνία για το Κακάο. Νομίζω ότι θα βοηθήσει ε, για την κοινωνική και περιβαλλοντική σταθερότητα εκεί ε, του κλάδου του κακάο. Αλλά ανησυχώ επίση βαθύτατα για την παιδική εργασία σε αυτό το κλάδο. Α είμαστε όμω σαφεί η ευθύνη δεν είναι ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε των καταναλωτών στην Ευρώπη αλλά του κλάδου του κακάου. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαν 700 δισεκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό είναι αυτό κέρδη. Και δαπάνησαν 0,075% ε, ε, επενδύοντας στις ε, συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Ο κλάδος θα πρέπει να μορφώσει τα παιδιά που εκμεταλλεύεται, να βελτιωθούν οι συνθήκε εργασία ε, στι φοιτίες και στα εργοστάσια για να προστατεύονται τα παιδιά. Τελικά, όπω σα είπα, εγώ καλωσορίζω την ε, συμφωνία και την έκθεση, αλλά για μα ο καλύτερο τρόπο να απαντήσουμε είναι να υποστηρίζουμε το δίκαιο εμπόριο και να αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα. Μάλιστα, παίρνουμε στο ΚΑΤΣΙΑΙ, κυρία Αντζελίλη, για ένα λεπτό. She's not για ένα λεπτό ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κακάο παράγεται σε 40 χώρες με 8 εκατομμύρια εκτάρια φυτιών. Όμως τελικά η παραγωγή αυτή επιφέρει μεγαλύτερη φτώχεια στις χώρες αυτές. Ο τομέας λοιπόν δεν δίνει απαραίτητο εισόδημα σε 50 εκατομμύρια ανθρώπων από τον κόσμο. Παρόλο που είναι βιοποριστικό τομέα, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νομικό σύστημα που θα προβλέπει δικαιότερου όρου για την εργασία των ανθρώπων αυτών, η παραγωγή, από, αλλά για όλη την αλυσίδα παραγωγή, από τον ε, καλλιεργητή μέχρι τον καταναλωτή. Το εμπόριο του προϊόντο αυτού θα πρέπει να βασίζεται λοιπόν σε δίκαιε προποθέσει και όρου και να γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές ε, και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Εδώ χρειάζονται δικαιότερες τιμές, γεγονός που θα βοηθούσε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που για να εδώ συζητήσαμε, όπως η παιδική εργασία. Για ένα λεπτό, η κυρία Μάιστερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η σοκολάτα και το κακάο δεν είναι κάτι που εφραίνει την καρδία των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Τώρα μπορεί να είμαστε στο Στρασβούργο, αλλά συνήθως είμαστε στις Βρυξέλλες και ε, ε, το σοκολατάκι και οι της Βρυξελών είναι κάτι που ο κόσμος αγοράζει ευχαρίστως και ε, προσφέρει κιόλα. Και δεν σκέφτεται πώς έχει παραχθεί το κακάο, ούτε τι έγινε στις φοιτήσεις, ούτε πώς γίνεται η σοκολάτα. Το καταλάβαμε όμως από τη συζήτηση ότι πρέπει να μας προβληματίσει αυτό, ότι συνδέεται με παιδική εργασία για να μπορέσουμε να εισαγάγουμε καν αυτό το κακάο. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό που είπε η κυρία Κέρστιγκερ, αν έχουν εκεί την οικογένειά τους ή αν τους καταναγκάζουν να δουλεύουν. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας, πώς δουλεύουν και ε, αυτό βλάπτει την υγεία τους. Είναι μαζικές οι ε, συνέπειες στην υγεία τους ε, για τον τρόπο με τον οποίο παράγεται καν το κακάο από παιδιά και από παιδιά. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε χώρες όπως η Γκάνα και η ακτή ελεφαντοστού, οι αναπτυσσόμενες χώρες που προσπαθούν έτσι να έχουν ε, ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους λαούς τους, να ε, έχουν συμμετοχή στο δίκαιο εμπόριο, το είπαν πολλοί. Και νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ειδικό σήμα για τη σήμανση αυτών των προϊόντων και θα ήταν μια καλή λύση. Και χαίρομαι για την ομοφωνία στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Επίτροπο, έχει το λόγο ο κύριο Πίμπαλξ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, Βλέπουμε νομίζω μια ευπρόσδεκτη σύγκληση απόψεων να εκδηλώνεται από αυτή τη συζήτηση. Είναι όντω ε, πολύ καλό προϊόν το κακάο. Επίση για πολλέ χώρε, και αν, αν λογιστείτε την ακτή ε, του ελεφαντοστού ω παράδειγμα, είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν ε, στην οικονομία του. Είναι πολύ σημαντικό εκ τούτου να έχουμε θεμητέ συνθήκε εμπορίου και καλέ τιμέ για την αγορά του προϊόντο. Ο κλάδο πρέπει να μεριμνά μόνο του ώστε να μην υπάρχει η αδίποτε σκιά στην, στις διαδικασίες παραγωγής και να είναι πάντοτε θεμητές οι συνθήκες παραγωγής. Και στην ε, συσκευασία επίσης, προσπάθειες που έχουμε ήδη κάνει με την Κάνα και την άκρη του Λεφαντοστού, αλλά και πολλά άλλα πράγματα που μένουν να γίνουν, και εν προκειμένου βέβαια το ζήτημα της εργασίας των παιδιών, όπως και άλλα. Και θα θέλω εδώ να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει διαδικασία ευαισθητοποίησης για την εφαρμογή της ε, συνθήκης ε, του οργανισμού Διεθνού Οργανισμού Εργασία υπαριθμών 182 για την απαγόρευση τη εργασία των παιδιών και τη συμβάσεω για, ε, για τα δικαιώματα του παιδιού. Η προστασία λοιπόν των παιδιών από την εργασία έχει αναγνωριστεί και καταγραφεί ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλές από τις στρατηγικές σε σχέση με χώρες που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με τους εμπορικούς μας εταίρους προάγουμε και τον πολιτικό διάλογο παράλληλα, όχι μόνο σε εμπορικές σχέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουν και την προτεραιότητα αυτά τα ίδια τα ενδιαφερόμενα κράτη. Έχει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδώσει αυτόν τον οδηγό για μια για ένα δημόσιο σύστημα δημοσίων ε, συμβάσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την παιδική εργασία, αντίστοιχα, προβλήματα, προγράμματα μάλλον για την ανάπτυξη που στόχο έχουν ενώ ξέρω να εξαλείψουν την παιδική εργασία. Φερρυπίν το πρόγραμμα Τάκλι με 40 εκατομμύρια ευρώ που απευθύνεται σε 14 χώρες ΑΚΕ και προτείνει λύσεις για την εκπαίδευση κατάρτιση παιδιών και πέρυσι ε, οι προτάσεις που είχαμε για την αντιμετώπιση της ε, εργασίας των παιδιών. Στο τομέα του κακάοδαντρου συγκεκριμένα έχουμε πρόγραμμα το οποίο έχει ουσιαστικά βελτιώσει την, ε, τα εισοδήματα, τα των εισοδημάτων των ε, γεωργών, στην Κάνα κυρίως, και έχει βελτιώσει συνθήκες παραγωγής εκεί. Σας βεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει πιστή στην επιταγή μιας, κοινωνικ... μιας πολιτικής συνοχής και συνέπειας ως προς τις εμπορικέ μας σχέσεις με την πραγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ευαισθησίας. Ε, το ζήτημα των τη εργασία των παιδιών όμω δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα και σε ένα χωριστό πρόβλημα. Οι εμπορικέ ε, σχέσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένε ε, διατάξεις εκ τούτου για την βελτίωση των συνδικών εργασία των εργαζομένων και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και την ειχνηλασιμότητα των προϊόντων εφόσον αυτά έχουν παραχθεί δηλαδή με παιδική εργασία πρέπει να το να τα εντοπίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτροπε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μαρέα. Ε, ε, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή, ιδιαίτερα στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τελικές συμβαστικές προτάσεις για το θέμα της καταπολέμησης της ε, παιδικής εργασίας είναι και ευπρόσδεκτα και εύστοχα. Εδώ θέλω να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιθυμούμε να πιστέψουμε σε αυτά που μα λένε. Πραγματικά εδώ χρειάζεται να υπάρξει απαραίτητη πολιτική βούληση για να κυρωθεί και να υλοποιηθεί σωστά ε, η σύμβαση του οργανισμού, Οργανισμού Εργασίας ε, κατά τη παιδική εργασία. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτή την κίνηση προκειμένου να έχουμε και κέρδη στην ε, διάσταση της βιωσιμότητας του, της αγοράς του κακάο και κυρίως θα πρέπει να διερευνήσουμε την όλη ιδέα της ιχνηλασιμότητας, ιχνηλασιμότητας ε, των προϊόντων κακάο ώστε να δημιουργηθεί ένα σήμα απαλλαγμένων από υποψίες εκμετάλλευσης παιδιών, παιδικής εργασίας για τα προϊόντα του κακάου. Αυτό θα ήταν το ο καλύτερο τρόπο ε, τη αναγνώρισε τη σημασία του όλου θέματος στην παραγωγή κακάου. Και ήθελα να προσθέσω και το εξή. Σε ό,τι αφορά τι διεθνεί εμπορικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι διεθνεί μα εμπορικέ συμφωνίε, το θέμα αυτό δεν μπορεί να μην περιλαμβάνεται. Θα πρέπει στι συμφωνίε τη εταιρική συνεργασία και σύνδεση με τι χώρε ΑΚΕ να λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο αυτό. Γιατί μιλάμε για χώρε που παράγουν κακάο. Δεν μπορεί να μην παραλαμβάνεται λοιπόν αυτό. Έχει μια ε, πανοπλία εμπορικών μέτρων λοιπόν, ένα εμπορικών μέσων στα χέρια της Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, μια διάσταση που ανέφερε και ο Επίτροπος ε, μέσω του συστήματος διαφοροποιημένων ε, προτιμήσεων. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να μην ξεχνάμε ότι οι ενδιαφερόμενοι πολλές φορές σε αυτό το τομέα είναι ευρωπαϊκές εταιρείε που και εκείνοι έχουν την ευθύνη τους στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτρο. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση λοιπόν. Κοινή συζήτηση για το τομέα του κακάου. Ένα σχέδιο ψηφίσματος έχει κατατεθεί ε, για τη ε, συζήτηση του θέματος αυτού. Είπα, μίλησε τελευταίος ο εισηγητής. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο ε, σημείο της ημερησίας διάταξης, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής